για να ξεκινήσουμε. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie. Άρχεται η συνεδρίαση. Ε, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου και με λύπη σας πληροφορώ πως η Πίλαρ Χουάρες Μποά, η υποδιευθύντρια της ε, αποστολής μας στην ΑΕΤ, εξακολουθεί να αγνοείται. Αναζητείτε ακόμα η Πίλαρ ήταν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, Σήμερα η σκέψη μας πηγαίνει στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή την ε, τραγωδία. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγγείλει πώς θα στείλουν σημαντική οικονομική βοήθεια και 150 αστυνομικούς μεταξύ άλλων. Πολλά κράτη-μέλη έστειλαν και ε, άλλη βοήθεια. Είναι, μια, είναι η σημαντικότερη καταστροφή στην ιστορία της ΑΕΤ και μία από τις ε, σημαντικότερες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αγνοούνται επίσης πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.